Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα ενώπιόν σας ως υποψήφιος για να αποτελέσω μέλος του επιτελείου του πρώτου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξελέγει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ε, βρίσκομαι μπροστά σας έχοντας περάσει 13 χρόνια στα έδρανα αυτά χρόνια που τα θεωρώ από τα καλύτερα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας και του πολιτικού μου βίου. Γνωρίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γνωρίζω ότι ανέκαθεν υπεράσπιζε το ευρωπαϊκό συμφέρον και τις ευρωπαϊκές αξίες. Τις οικουμενικές αξίες της δημοκρατίας, ελευθερίας, δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και ισότητας που είναι τα θεμέλια που έκαναν την Ευρωπαϊκή Ένωση από τι πιο ευημερούσε και ελεύθερε περιοχέ του πλανήτη. Είναι αξίε που μα ενώνουν ω δημοκράτε και Ευρωπαίου και διαπότιζαν ανέκαθεν την πολιτική μου δράση και αυτό θα κάνω και στο μέλλον. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην αρχή τη ισότητα. Στην προεκλογική εκστρατεία που πέρασε, έκανα ένα ατυχέ σχόλιο που έθεσε ένα αμφιβόλο τη δέσμευσή μου υπέρ τη αξία τη ισότητα. Ήταν όντω ένα ατυχέ σχόλιο. Ζήτησα συγγνώμη και τότε και θα ήθελα και πάλι να ζητήσω συγγνώμη. Λυπάμαι. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι σημαντικός ακρογωνιαίος λίθος ε, για να δημιουργήσουμε μια πιο δίκαιη, πιο ευημερούσα και, πιο, ε, και μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω κάποιες πληροφορίες που κυκλοφόρησα τις τελευταίες μέρες. Δεν πραγματοποίησα καμία απολύτως αλλαγή στη δήλωση οικονομικών μου συμφερόντων ε, ως επίτροπος. Και όλες μου οι δραστηριότητες και οι επαγγελματικές και οι πολιτικές αντικατοπτρίζονται πιστά στη δήλωση αυτή. Σε ό,τι αφορά το πόθεν έσχεση του Ευρωβουλευτή, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι χθες έκανα την ενημέρωση της δήλωσης αυτής μετά από αλλαγή των περιστάσεων που αναφερόταν στην δήλωση αυτή. Ήθελα να συμπεριλάβω την ολοκλήρωση της πώληση των μετόχων των εταιριών Πετροκλής και του ΚΑΡ, όπως είχα προαναγγείλει. Ούτε εγώ, ούτε κανένα από το στενό οικογενειακό μου κύκλο δεν έχουμε κανένα δεσμό με τι επιχειρήσει αυτέ. Και μάλιστα από αυτή την άποψη πήγα πολύ πιο μακριά από τι απαιτήσει τη ισχύουσα νομοθεσία. Επίση, θα ήθελα να σα ενημερώσω για την παρέτησή μου από τη θέση του Προέδρου του Ιδρύματο ΦΑΕΣ μετά την, τον ορισμό, το διορισμό μου ω υποψηφίου επιτρόπου. Και επίση, συμπεριέλαβα στο, στη δήλωσή μου και το αξίωμα του Προέδρου τη Εθνική Εκλογική Επιτροπή του Κομματό μου από το 2008 μέχρι το 2011. Αυτό το αξίωμα περιλαμβανόταν και στη δήλωση ε, συμφερόντων που υπέβαλα στην Επιτροπή και στο βιογραφικό που υπέβαλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα νευραλγικό σημείο της δημοκρατικής ζωής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είμαι υπέρ ενός ε, σημαντικού διαλόγου μαζί του που θα αποτελέσει τη βάση οποιασδήποτε πρόταση θα υποβάλω. Είμαι στη διάθεσή σας και πρόθυμος και εγώ και οι υπηρεσίες μου για να έρθω για διάλογο, εξηγήσει ε, και για να ακούσω τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο διάλογος μας βοήθησε να ξεπεράσουμε εθνικούς εγωισμούς υπέρ ενός κοινού σχεδίου αλληλεγγύης που αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μεγάλη αίσθηση ευθύνη αναλαμβάνω την ε, δέχομαι την πρόταση που μου έγινε για να λάβω την, το χαρτοφυλάκιο των κλιματικών αλλαγών και της ενέργειας. Οι δύο πολιτικές αυτές είναι πολύ σημαντικές και θα σημαδέψουν το πεπρωμένο των επερχόμενων γενεών. Έχω ακράδαντες πεπιθήσεις, πιστεύω ότι θα πρέπει να πρωτοστατήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έτσι θα εξασφαλίσουμε και την ανταγωνιστικότητά μας και θα δημιουργήσουμε και θέσεις απασχόλησης. Και φυσικά οι προσπάθειές μας θα πρέπει να έχουν μια διαχρονικότητα και να είναι και αποτελεσματικές και να έχουν και απτά αποτελέσματα. Πιστέψτε με, από την πολιτική μου πείρα ως υπουργό Περιβάλλοντος είχα πολύ αποφασιστική και ξεκάθαρη δράση ε, και στήριξα τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα των κλιματικών αλλαγών. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να πρωτοστατήσουμε στη, μάχη, στη μάχη αυτή. Συνεργάστηκα στενά με την Επίτροπο Κόνι Χέντεγκαρτ και θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή στο έργο της και στους συνεργάτες της. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε θαραλέοι και φιλόδοξοι σε αυτές τις πολιτικές. Κατά τη γνώμη μου, η απόφαση να συνδεθούν οι κλιματικές αλλαγές και η ενέργεια είναι ένα σημαντικό μήνυμα που θέλει να δώσει για τις πολιτικές αυτές ο εκλεγμένος πρόεδρος Γιούγκερ. Θέλουμε μια φιλόδοξη πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές και μια ενεργειακή πολιτική με βιώσιμο χαρακτήρα. Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και μάλιστα είναι σημαντικό που και τα δύο αυτά θέματα εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο του ίδιου επιτρόπου. Έτσι θα εξασφαλίσουμε συνοχή των πολιτικών και θα δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνέργειες για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και ισχυροί. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα πλαίσιο για το 2030 για το κλίμα και την ενέργεια αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το θετικό χαρακτήρα αυτής της ολοκληρωμένης εστίασης. Η προκλήσεις είναι πολλαπλές. Θα πρέπει με αποφασιστικό τρόπο να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, να μειώσουμε την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, να δημιουργήσουμε ένα ενεργειακό σύστημα που θα εξασφαλίζει ενέργεια σε προσιτές τιμές για όλους τους καταναλωτές, να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού, να μειώσουμε την ε, εξάρτησή μας από τις εισαγωγές και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Και όλα αυτά θα τα επιτύχουμε αν συνενώσουμε τις προσπάθειά μας και δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο. Έχουμε τεράστιο δυναμικό. Η εντολή που ανέλαβα από τον εκλεγμένο πρόεδρο είναι σαφής. Είναι καταρχήν σημαντικό να διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στην Σύνοδο Κορυφής για το Περιβάλλον των Παρισίων του 2015. Γι' αυτό και θα ήθελα να επισημάνω το, τη σημασία να είναι, να είναι φιλόδοξο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου και σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρόκειται για μια συλλογική ευθύνη που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Θα πρέπει να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνιστής ε, σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών αλλά και για βιώσιμες θέσεις ανάπτυξης. Θα ήθελα ο κόσμος να συνδέει, να κάνει το συνειρμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την Ευρώπη. Θέλουμε φυσικά και δίκτυα που θα είναι ε, σύγχρονα και θα μπορούν να εκμεταλλεύονται στο έπακρο το δυναμικό αυτών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέλουμε να γίνει η Ευρώπη ε, η πιο αποδοτική ήπειρο σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργεια. Ήταν σαφή ο πρόεδρο Γιούγκερ. 30% υποχρεωτική ε, ενεργειακή απόδοση για το 2030. Απαραίτητη προπόθεση. Και θα συνεργαστώ μαζί σα για να προωθήσουμε τι απαραίτητε πολιτικέ, ε, επιδιώκοντα φυσικά τη συνένεση. Όλα αυτά θα γίνουν λαμβάνοντα υπόψη ότι η δημιουργία μια στιβαρή ενεργειακή ένωση και μια διορατική πολιτική για τι κλιματικέ αλλαγέ θα αποτελέσουν σημεία κλειδιά για το μέλλον. Διανύουμε τεραγμένου καιρού και η όλο και μεγαλύτερη αστάθεια στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δημιουργούν ε, προβλήματα και έχουν συγκεκριμένε συνέπειε. Γι' αυτό ύψιστη προτεραιότητά μου θα είναι η εξασφάλιση του ενεργειακού ε, ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο τον, οκτώ, τον, το φθινόπωρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου ο Επίτροπος Έντιγκερ υπέβαλε πρόταση για συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για να αποφευθούν προβλήματα στον ανεφοδιασμό σε φυσικό αέριο το φθινόπωρο. Εγώ πιστεύω στη διπλωματία και θεωρώ ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η λογική για να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου όλοι θα βγούμε χαμένοι. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστώ ε, άοκνα. Η τροτότητα της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την ενεργειακή εξάρτηση είναι γνωστή. Γι' αυτό και η ενεργειακή ασφάλεια θα πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα. Και από αυτή την άποψη, ω Επίτροπο Κλιματικών Αλλαγών και Ενέργεια, θα συμβάλλω υπό το συντονισμό τη Αντιπροέδρου για την, ε, για την Ενεργειακή Ένωση θα συμβάλλω στην δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενέργειας με μια φιλόδοξη πολιτική κλιματικών αλλαγών που θα στηρίζεται στους ακόλουθους πυλώνες. Καταρχήν, μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση πέρα το 2020, κυρίως ε, στα, στα κτίρια, στις μεταφορές και σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Επίσης θέλουμε μια ουσιαστική ενιαία αγορά της ενέργειας με ελεύθερη κυκλοφορία της. Γι' αυτό Χρειαζόμαστε διασυνδέσεις και δίκτυα απόλυτα ολοκληρωμένα μεταξύ τους και να θέσουμε ένα τέρμα στις ενεργειακές νησίδες, είτε είναι φυσικές είτε κανονιστικές, βάζοντας τους καταναλωτές στην καρδιά και το επίκεντρο των αποφάσεών μας. Θα πρέπει να μειώσουμε την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας νέες πηγές και διαδρομές εισαγωγής. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη διαπραγματευτική μας δύναμη και να χρησιμοποιήσουμε αμφίδρομες ροές ενέργειας. Γι' αυτό και το γρήγορο άνοιγμα του νοτίου διαδρόμου θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο της ενεργειακής πολιτικής υπέρ της διαφοροποίησης και της ενεργειακής ασφάλειας. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε την, την τεχνολογική ανάπτυξη και την έρευνα σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες θα πρέπει να εφαρμόσουμε νέες τεχνολογίες με χαμηλή χρήση άνθρακα που θα είναι αποδοτικές ενεργειακά. Επίσης θα πρέπει να αυξήσουμε και την δική μας παραγωγή ενέργειας και να βελτιώσουμε το συντονισμό των εθνικών ενεργειακών πολιτικών προκειμένου ε, να είμαστε ενωμένοι απέναντι στις τρίτες χώρες. Χρειαζόμαστε και ένα νέο σύστημα κοινή ενεργειακή διακυβέρνηση, για να εξασφαλίσουμε μια πραγματική κουλτούρα ενεργειακή συνεργασία και σε περιφερειακό επίπεδο. Θα ήθελα να υλοποιήσουμε πλήρως το πλαίσιο του 2030, συνδυάζοντα όλους τους μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας. Και γι' αυτό θα σας υποβάλω για κάποιες ιδέες. Θα ήθελα να ενισχυθεί το σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Προτεραιότητά μου είναι η έγκριση του αποθεματικού σταθερότητα τη αγορά για να εξασφαλιστεί η διαρθρωτική σταθερότητα που χρειάζεται η αγορά του άνθρακα. Και επίση θέλω να ενισχυθεί αυτό το σύστημα για να εξασφαλίσουμε συμμόρφωση με του κλιματικού στόχου μετά το 2006 με αποδοτικό και ε, προσοδοφόρο τρόπο. Επίση, μετά από ένα πολιτικό διάλογο μαζί σα, θα υποβάλω νομοθετική πρόταση προκειμένου η κατανομή των εκπομπών αερίου του θερμοκήπιου που δεν ανακαλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών να κατανεμηθούν μεταξύ όλων των τομέων. Σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, θα χρειαστούμε προσαρμογή και σταδιακή μετατροπή όλων των συστημάτων προκειμένου να βρεθούν οι απαραίτητες ισορροπίες. Και τέλος, θέλουμε μια μετάβαση σε μια οικονομία που θα χρησιμοποιεί πολύ λιγότερο άνθρακα και που θα πρέπει να συνδυάζεται με την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και την καινοτομία. Θα πρέπει ταυτόχρονα να καταπολεμήσουμε την ανεργία, ιδιαίτερα των νέων. Και από αυτή την άποψη ο πρόεδρος Γιούκερ θα υποβάλει μια πρόταση, ένα πακέτο για την απασχόληση με επενδύσεις που θα έρθουν σε 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλουμε αυτά αποτελέσματα ώστε οι κλιματικές αλλαγές και η ενέργεια να αποτελέσουν προτεραιότητα και της μελλοντικής αυτής πρότασης και του πακέτου. Αυτό προποθέτει βέβαια συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και πολύ διάλογο. Η ενέργεια και το κλίμα δεν έχουν πολιτικά χρώματα. Ούτε είναι σε αντιπαλότητα μεταξύ του. Θα πρέπει να κάνουμε μια συλλογική προσπάθεια. Ούτε ένα άνθρωπο στον πλανήτη δεν θα μείνει στο απειρόβλητο των κλιματικών αλλαγών. Ούτε μια γωνιά στην Ευρώπη. Ούτε ένα σπίτι. Ούτε μια επιχείρηση δεν θα απαλλαγεί από τι συνέπειε και μάλιστα θα ζήσει τι συνέπειε και από ενεργειακή άποψη. Ε, δεν μπορούμε να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Το διακύβευμα είναι τεράστιο και για να ανταπεξέλθουμε από κοινού στη μείζον αυτή πρόκληση ζητώ την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ.